15-16 για την επικορικότητα και την αναλογικότητα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εδώ και πολλά χρόνια είμαι εισηγήτη όσον αφορά την ετήσια έκθεση για την αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας και όλο και περισσότερο με ικανοποιεί αυτό το θέμα. Εκτός του ότι είναι το τελευταίο θέμα στην Ολομέλεια στις 10 και Θέλω να υπενθυμίσω ότι οι αρχές αυτές δεν είναι μια έκκληση για δράνεια, αλλά κανόνες κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κρατών μελών. Ε, λοιπόν, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός αν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα, δεν μπορεί να παρεμβαίνει παρά μόνο σε θέση να δράσει αποτελεσματικότερα από ό,τι τα κράτη-μέλη σε εθνική ή τοπική κλίμακα. Το ίδιο η αρχή της αναλογικότητας προβλέπει ότι τα μέσα που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση στόχων που καθορίζουν οι συνθήκες δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα αναγκαίο. Αυτές οι αρχές θεωρήθηκαν ότι εγγυούνται την αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσης. είναι και βασικά μέσα για τη σχέση Ευρωπαϊκής Ενώσης με τους πολίτες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιούνται για δημιουργία προβλημάτων, κολυσιεργίας ή να τροφοδοτούν τον ευρωσκεπτικισμό. Το αντίθετο, μάλιστα. Η παρούσα έκθεση καλύπτει τα έτη 2015 και 2016 και διατείνεται ότι τα εφιστάμενα μέσα ε, είναι πολλά μια πανοπλία εργαλείων που επιτρέπει τη συμμετοχή στα διάφορα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μελέτης αντικτύπου, δημόσιες διαβουλεύσεις, η πλατφόρμα REFIT, η πλατφόρμα IPAX, η πλατφόρμα εσωτερική RECPAX και CONNECT. Ο διάλογος ε, μέσω COSAC και Επιτροπής των Περιφερειών, χωρίς να συσμονούμε, τη διαδικασία της ε, κίτρινης κάρτας ε, και από το 2014 τα Εθνικά Κοινοβούλια εκδήλωσαν αυξημένο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή πολιτική μέσω των νέων εργαλείων που δημιουργήθηκαν κυρίως μέσω του REFIT. Το 2016-65 γνωμοδοτήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων παρελήθησαν μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2015 και είναι κάτι ενθαρρυντικό. Άρα δεν είμαι υπέρ ε, και δημιουργίας νέων μέσων χωρίς να διαρευνηθεί πλήρως το δυναμικό των υφισταμένων εργαλείων. Η διαδικασία λειτουργεί όταν όλοι οι πρωταγωνιστές ε, ε, ενδιαφέρονται γι' αυτό. Υπογραμμίζω ότι δεν χρειάζεται να δημιουργούμε νέες διαδικασίες και εργαλεία που θα, επιφόρτωναν, θα επιφόρτωναν μάλλον ε, τις διάφορες διαδικασίες και θα παρεμπόδιζαν την νομοθετική διαδικασία. Πιστεύω ότι μαζί, μαζί με τους Κιώδης κατορθώσαμε να ετοιμάσουμε ισορροπημένη έκθεση που ζητά να έχουμε μια αποτελεσματική ένωση που θα ακούει τους πολίτες και θα σέβεται τη διαφορά και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την συνεργασία τους και ήταν πολύ ευχάριστη συνεργασία. Τέλος, όσον αφορά την Task Force Timmermans, όπως αποκαλείται, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ δημιούργησε μια μάδα εργασίας που είναι επιφορτισμένη με τον προβληματισμό ε, επί της επικουρικότητας. Εκλήθησαν εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων, τη Επιτροπή των Περιφερειών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η άρνηση του Ευρωκοινοβουλίου να συμμετάσχει ε, δεν εκφράζει έλλειψη ενδιαφέροντο από πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου, κατά την άποψή μου, αλλά ε, ζητά να σεβασ... γίνει σεβαστός ο ρόλος του συνομοθέτη. Και οι ευρωβουλευτές έχουν κάθε δυνατότητα να εκφραστούν εκ των υστέρων όσον αφορά τα αποτελέσματα των εργασιών της Task Force. Αυτή η απουσία του Ευρωκοινοβουλίου δεν θα πρέπει επουδενή να επιδεινώ στη σχέση του Ευρωκοινοβουλίου με την Κόσα και την Επιτροπή των Περιφερειών. Θα ήθελα οι σχέσει μα με την Επιτροπή των Περιφερειών να ενισχυθεί και έγραψε επιστολή εν αυτή τη ενία απευθυνόμενη προ τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα θεσμό απαραίτητο διότι αποτελεί έναν ομφάλιο λόρο που συνδέει τι περιφέρειες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται προσέγγιση λοιπόν μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, εθνικών τέτοιων φορέων και τοπικών. Μόνο μαζί καθένα στην κλίμακά του μπορούμε να δράσουμε και να εφαρμόσουμε μια πολιτική που είναι ε, η αναγκαία για την ευημερία των πολιτών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Ντελβό. Το λόγο έχει ο κύριος Μίμητσα. Thank you, Madam Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Τελβό για την εξαιρετική δουλειά που έκανε και τα θετικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει. Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της, η Επιτροπή Γιούνκερ προσπάθησε να δώσει σάρκα και οστά και να εφαρμόσει πλήρως τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Θέλουμε να συνεργαζόμαστε με τα Εθνικά Κοινοβούλια και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις αρχές αυτές. Γι' αυτό και λοιπόν με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσουμε την κατανόησή μας ως προς το τι σημαίνει επικουρικότητα και αναλογικότητα. Οι διοργανικές συμφωνίες για καλύτερη νομοθεσία που υπέγραψαν τα τρία θεσμικά όργανα πρόσφατα δίνουν έμφαση στην διασφάλιση του σεβασμού αυτών των αρχών, στην νομοθεσία και στην αξιολόγηση του αντικτύπου αυτής. Φαίνεται η κοινή δέσμευση για να επέλθει αυτή η αλλαγή που θέλουν να δουν οι πολίτες στην Ευρώπη. Ο συνάδελφός μου, ο αγαπητός κύριος Φρανς Τίμερμανς, θα ήθελε πολύ να είναι εδώ απόψε, όμως έπρεπε να μεταβεί στο Λουξεμβούργο για το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Υπό την ηγεσία του, το Σώμα των Επιτρόπων έχει ε, δώσει μεγάλη έμφαση στην καλύτερη νομοθεσία και έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη ε, συμμετοχή των πολιτών και ε, διαμόρφωση κανόνων βασισμένων σε στοιχεία. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά και πάνω σε αυτά ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην ε, δήλωσή του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017 ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε μια task force για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα με στόχο να ε, βελτιωθεί η εφαρμογή το Νοέμβριο του 2017 έγινε αυτό. Αυτό πρέπει να λαμβάνει χώρα στο κατάλληλο επίπεδο, είτε αυτό είναι ευρωπαϊκό, είτε τοπικό, είτε περιφερειακό. Όπου υπάρχουν τομείς πολιτικής που θα μπορούσαν οι αρμοδιότητες να ε, περάσουν πάλι στα κράτη-μέλη ή στις περιφέρειες, αυτό ε, είναι το επιθυμητό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει επίσης ότι οι έδρες για το η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραμένει διαθέσιμη. Αυτό που συζητάμε σήμερα, η έκθεση δηλαδή αυτή, δείχνει το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, εφαρμογή και τον έλεγχο της εφαρμογής της αρχής της επικουρικότητας. Αυτή τη στιγμή η Task Force εξετάζει παρόμοιες προτάσεις με αυτές που περιέχει η έκθεση. Ο έλεγχος της επικουρικότητας έχει έναν ε, μηχανισμό για το σκοπό αυτό και θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας ε, εκθέσει τους λόγους για τους οποίους νομίζει πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σέβεται την αρχή της επικουρικότητας. Ζητήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ενημερώνει το Κοινοβούλιο για τις αιτιολογημένες γνώμες που λαμβάνει από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτές είναι ήδη δημοσιευμένες στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, η εξαίρεση των περιόδων διακοπή, διακοπών, ε, όπως ε, τον Αύγουστο, ζητήθηκε να είναι 8 εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή η Task Force εξετάζει τα θέματα αυτά και τη σχέση τους με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Ε, τέλος να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει το μονοπόλιο στις ε, καλές προτάσεις. Πάντα είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε προτάσεις και ιδέες από τα Εθνικά Κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2015 υπήρξε μια πρωτοβουλία για ε, τη σπατάλη τροφίμων στα πλαίσια της πράσινης κάρτας και πολλοί ε, εξέτασαν το, την αντίστοιχη δέσμη μέτρων που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015. Συμφωνώ μαζί σας με το ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δείχνουν πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην διαδικασία αυτή θεωρούμε πως έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ε, χρησιμοποίηση των υφιστάμενων ε, μηχανισμών ε, στο σύνολό τους και στο όρο των δυνατοτήτων τους παρά να δημιουργήσουμε νέα μέσα που θα χρειαστούν αλλαγή των συνθήκων. Αυτά από μένα σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ντελβό για τη σύνταξη της έκθεσης αυτής ε, και ευχαριστώ και επιθετήσατε πολλές προτάσεις της ΕΦΚΟ. Υπάρχει συμφωνία ότι οι αιτήσει εκθέσει για επικουρικότητα και αναλογικότητα είναι πολύ σημαντικά εργαλεία για να ε, διατηρήσουμε τα προνόμια των Εθνικών Κοινοβουλίων που αναγνωρίζεται από τη συνθήκη. Επίση, για να μπορούμε ε, να δούμε ότι η επικουρικότητα και η αναλογικότητα λειτουργούν ε, σωστά. Το βλέπουμε ότι υπάρχει ένας μικρός αριθμός κίτρινων καρτών ε, που έχουν υιοθετηθεί σε ό,τι αφορά τις ετυλογημένες γνώμες των Εθνικών Κοινοβουλίων. Στο, έχει γίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένας ε, εταίρος που συμμετέχει ενεργά στο διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια. Πρέπει να υπάρχει μια δόση ευελιξία στο σύστημα έγκυρης προειδοποίησης στην ε, ερμηνεία των προθεσμιών ε, και θα πρέπει να υπάρξουν και λεπτομέρειες σε σχέση με την υλοποίηση των διατάξεων που αναφέρονται στις συνθήκες για τα εθνικά κοινοβούλια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο κύριος Ράντεφ για το ΕΛ και για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να συγχαρώ το, την εισηγήτρια και να την ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας για την καλή συνεργασία που είχαμε όσον αφορά αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους άλλους κοιόδης εισηγητές. Ε, νομίζω ότι αυτή η έκθεση πετυχαίνει τη σωστή ισορροπία, αντικατοπτρίζει επακριβώς τα βασικά σημεία τη ετησία εκθέσεω Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επικουρικότητα και αναλογικότητα για το 2015 και 2016. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι πρωτοβουλίε που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια και που συνέβαλαν στην σωστή εφαρμογή των δύο αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση κρίση ανεκπροηγουμένου και προσπαθεί να βρει την ταυτότητά της, είναι αρκετά σημαντικό να υπάρχει μια στέρεη ευρωπαϊκή νομοθεσία στους τομείς όπου η Ένωση μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά και να δώσει προστιθέμενη αξία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να εφαρμόζουμε επακριβώς τις δύο αρχές. Αν δεν το κάνουμε αυτό θα δώσουμε μόνο φωνή στους ευρωσκεπτικιστές. Τα εθνικά κοινοβουλία εκπροσωπούν τους Ευρωπαίους πολίτες σε εθνικό πλαίσιο. Είναι αρκετά σημαντικά τα εθνικά κοινοβούλια για να ξεπερνιόνται διαφορές απόψεων μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και του κοινού. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε πραγματική ευκαιρία να συμμετέχουν προβλέποντας μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον υπολογισμό της περίοδου των 8 εβδομάδων Εντό τη οποία περίοδου μπορούν να στείλουν την αιτιολογημένη του γνωμοδότηση. Εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας και της επικορικότητας, θα θεσπίζουμε καλύτερους κανόνες που δεν θα επικρίνονται. Μόνο έτσι θα μπορούμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εν ονόματι των Σοσιαλιστών, ο κ. Κονφεράτη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Η έκθεση που συζητούμε είναι έκθεση πάρα πολύ ισορροπημένη ε, και αυτό λόγω του πάθους που ε, διέθεσε ο συνάδελφος Τελβό για τη σύνταξη εκθέσεως. Το μέσο αυτό της ετήσιας εκθέσεως για θέματα επικουρικότητας και αναλογικότητας είναι σημαντικό εργαλείο, επιτρέπει να δώσουμε ουσία, σάρκα και οστά στην πρακτική που ακολουθούμε δημοκρατική, εξυπηρετεί την Ένωση. Η Ένωση χρειάζεται κάποιου τομεί να αναπτύξει και να διαδώσει τη νομοθεσία ε, μέσω πιο εντατική θέσπιση νομοθεσία και θα πρέπει να διοργανώνει την ήδη φυστάμενη νομοθεσία. Θα πρέπει να δώσουμε ένα σημαντικό μήνυμα, θετικό μήνυμα. Ε, θα το κάνουμε αυτό. Αν το καταφέρουμε αυτό, θέλουμε να το στείλουμε προ αυτού που μα κοιτούν, προ του Ευρωπαίου πολίτε θα στείλουμε το μήνυμα. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε ε, προ τα αιτήματα κάτωθεν και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι προτάσει και τα αιτήματα που προέρχονται από τα εθνικά κοινοβούλια ε, όπως αποκαλούνται ε, τα κίτρινες κάρτες. Ε, θα ήθελα επ' αυτού να δώσω ένα παράδειγμα. Το 2019 εννέα κοινοβούλια κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου για να εφαρμοστούν οι αρχέ τη κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Και εγώ ανανεώνω αυτό το αίτημα. Θα ήταν ένα καλό τρόπο για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε μια απέτηση που επιβεβαιώθηκε από σημαντικό αριθμό αιτήσεων που κατέφθασαν από αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καρίμ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό για το ECR. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ελπίζω να με ανεκτείτε, ενώ θα κάνω κάποια γενικά σχόλια και κάποια προσωπικά σχόλια. Καταρχήν ευχαριστώ τη Μάντη που έκανε αυτή την ε, τρομερή δουλειά εκ μέρου τη Επιτροπή μα και του Κοινοβουλίου. Αλλά θέλω να σε ευχαριστήσω επειδή ακού πάντοτε τι ε, προτάσει ε, που παρουσίασα. Δεν συμφωνούσε πάντα, αλλά ε, σε ευχαριστώ τουλάχιστον που ήσουν ανοιχτή στι ιδέε που πρότεινα για πολλά χρόνια. Εγώ ε, ασχολούμαι με το θέμα της επικουρικότητας και της αναλογικότητας ε, εκ μέρους ε, της Επιτροπής ε, και ε, φυσικά όταν παρουσιάζαμε αυτό το θέμα στο Κοινοβούλιο πάντοτε είχαμε ένα δείγμα δύναμης. Υπήρχαν κάποια θέματα όμως που δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου αυτή τη φορά. Παρ' όλα αυτά δεν θα καταψηφίσω την έκθεση γιατί είμαστε εδώ που είμαστε η θέση μου ήταν πάντα ότι θα πρέπει να δεσμεύσουμε, ε, να προσδέσουμε τα Εθνικά Κοινοβούλια στι διαδικασίε λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά, φτάνουμε στην κατάσταση που είναι η χώρα μου σήμερα και αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχω για να απευθυνθώ στο Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Καταλήγουμε σε μια Ευρώπη à la carte, ε, δηλαδή ότι ε, ουσιαστικά βρίσκει απήχηση στο λαό, το παρουσιάζουν οι κυβερνήσει ω δικό του έργο και ε, ότι προκαλεί δυσαρέσκεια το καταλογίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει όμως ε, να λογοδοτούν και τα εθνικά κοινοβούλια. Ευχαριστώ η κυρία Μπουτονέ για το ΕΝΕΦ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Καταρχήν, δεν μπορώ παρά να διαπιστώσω μια αλλαγή προς το καλύτερο στο ύφος και το περιεχόμενο αυτής της πρότασης για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα σε σχέση με το παρελθόν. Επίσης, ε, επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι ε, από τις ε, εκλογές και μετά θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε την επικουρικότητα και την αλογικότητα με ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ θα συνεχίσω βέβαια να επαγρυπνώ σε ό,τι αφορά την πραγματική εφαρμογή από τα ευρωπαϊκά όργανα αυτή της θεμελιώδη αρχή. Δεύτερον, χαιρετίζω ε, στο ότι τα Εθνικά Κοινοβουλία όλο ένα και περισσότερο χρησιμοποιούν την δυνατότητα που προβλέπεται από το πρωτόκολλο υπαριθμών 2. Ε, υποστηρίζω το να δημιουργηθεί μια διαδικασία κόκκινη κάρτας. Επίσης, η δυνατότητα να κατατεθεί αιτιολογημένη γνώμη θα πρέπει ε, να ε, καλύπτει όλη την ε, νομοθετική θητεία. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς τα Εθνικά Κοινοβουλία είναι η πραγματική δημοκρατική καρδιά της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ για το ΚΑΤΣΔΙ. Έχουμε και πάλι τον κύριο Μαριά, του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ένα λάθος ε, έκανα, μάλλον είναι επειδή είναι περασμένη ώρα. Ο κύριος ε, Πόσπισιλ επίσης είχε ζητήσει το λόγο. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Πόσπισιλ και μετά σε εσά, κύριε Μαριά. Μικρόφωνο για τον ομιλητή, παρακαλούμε. Ευχαριστώ. Ναι, Πάντοτε με ενδιαφέρει το θέμα τη αναλογικότητα και τη επικουρικότητα. Χαίρομαι που συζητάμε το θέμα αυτό εδώ. Δυστυχώς είναι αργά, μια περασμένη ώρα και δεν προσδίδεται η απαραίτητη προσοχή στην έκθεση αυτή, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτές οι δύο αρχές είναι απολύτως ζωτικές σε ό,τι αφορά την, ε, το νομοθετικό έργο. Χαίρομαι που βλέπω ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια πλέον ε, μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν ε, αυτό το εργαλείο της οτιολογημένης γνώμης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι στο μέλλον θα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο αυτά τα εργαλεία. Αυτό θα μας βοηθήσει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβαίνουν πράγματα ε, ε, δηλαδή του τύπου ε, οι εθνικοί νομοθέτες ε, να κάνουν δηλώσεις αν το ξέρουμε νωρίτερα ότι τέτοια νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήμασταν κατά. Εγώ υπερασπίζω τον κύριο Γιούνκερ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να έχουμε λιγότερη νομοθεσία αλλά καλύτερης ποιότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η έκθεση για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική. επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγκύτερα στους πολίτες. αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για μια αρχή δημοκρατική για μια αρχή η οποία οδηγεί σε αποκέντρωση εξουσιών και αυτό σημαίνει ότι επιλέγονται τα επίπεδα στα οποία θα λαμβάνονται οι αποφάσεις όταν πρόκειται για θέματα που εμπίπτουν σε αυτό που ονομάζουμε συντρέχουσες αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής ένωσης concurrent powers στα αγγλικά. άρα λοιπόν πρόκειται για ένα μηχανισμό ουσιαστικά νομιμοποίησης του ίδιου του ευρωπαϊκού εγχειρήματος καθώς δίνει πολύ σημαντικό ρόλο και στα εθνικά κοινοβούλια τα οποία διατηρούν ένα δικαίωμα βέτο ένα δικαίωμα της κίτρινης κάρτας να αμφισβητήσουν την δυνατότητα των βρυξελών να αποφασίζουν για όλα θεωρώ λοιπόν ότι στο βαθμό που λειτουργήσει η αρχή της επικουρικότητας σωστά εμπεδώνεται η δημοκρατία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης. ευχαριστώ. Κύριε Μιμίτσα, θα επανέλθουμε σε εσάς για τελευταία φορά απόψε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Mm. Τι, ε, τι θέλετε, κύριε Μπροκ. Εκτός μικροφώνου, ο κύριος Μπροκ. Ναι, ζήτησα να μιλήσω στα πλαίσια της διακασίας Catch the Eye τρεις φορές. Συγγνώμη, δεν με είδατε. Με αγνοήσατε. Λυπάμαι γι' αυτό. Μην λέτε τέτοια πράγματα κύριε Μπρόκ. Λυπούμε, δεν σα εντόπισα. Πραγματικά σα είδα για το Catch the Eye. Πραγματικά δεν σα είδα ότι ζητούσατε το λόγο για το Catch the Eye. Ζητώ συγγνώμη, λυπάμαι. Θέλετε κάπως αυτό να το αποκαταστήσουμε, να... Ναι, εάν ε, μου δώσουν αυτό το δικαίωμα να μου κάνουν αυτή τη χάρη, τρεις κυρίες, ναι, παρακαλώ, ε, σας ακούμε. Έχετε ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω αυτά τα δύο λόγια. Πιστεύω πως οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας είναι αποφασιστική σημασία και για ε, τα έθνη αλλά και για τις ίδιες τις αποφάσεις, διότι είναι ένα σημαντικό μέσο νομιμοποίησης Χρειάζεται όμως ταυτόχρονα να δούμε ότι αυτές οι δύο αρχές έχουν και μία αδελφή αρχή, την αρχή της αλληλεγγύης. Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα τρία, διότι κάποιες ε, χρόνες, χώρες ε, δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην επικουρικότητα και κάποιες ε, μικρότερες όχι, κάποιες πλουσιότερες ναι, κάποιες φτωχότερες όχι. Η αλληλεγγύη είναι πιο σημαντική για αυτέ. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να φροντίζουμε να μην γέρνει κάπου η πλάστιγκα. Όλοι έχουν το δικό του ρόλο. Έγινε λόγο για την κίτρινη κάρτα, υπάρχει όμω και η πορτοκαλή κάρτα στο πλαίσιο της συνθήκη τη Λισαβόνα, η οποία δεν πρέπει να παραμερίζεται και πρέπει να ενισχυθεί ο ε, ρόλος της, έτσι κι αλλιώς είναι πιο σημαντική από την κίτρινη κάρτα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πάντα να φροντίζουμε οι αποφάσεις να λαμβάνονται στο επίπεδο το οποίο προβλέπουν οι συνθήκες βάσει της αρμοδιότητας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπρόκ. Κύριε Μίμητσα, λυπάμαι που σας ε, καθυστέρησα. Έχετε τώρα το λόγο. Ευχαριστώ εκ νέου κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη να κλείσω διαβεβαιώνοντας όλα τα μέλη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει ούτω ώστε η αναλογικότητα και επικουρικότητα να παραμείνουν στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής Διαδικασίας και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μαζί σας, μαζί με το Συμβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, να κινηθούμε από αυτών και άλλων σημαντικών ζητημάτων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας ε, αξιότιμα μέλη. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η κυρία Ντελβό για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση ολοκληρώνεται όμορφα. Ακόμα και αν υπάρχουν αποχρώσεις ερμηνεών, νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη σύγκληση απόψεων επί της επικορικότητας, αναλογικότητας, ότι είναι σημαντικές αρχές. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπροκ που υπογράμμισε ότι η ε, ε, ε, βασική αρχή της λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η αλληλεγγύη που είναι μια αρχή που έχει και αυτή τη θέση της στο όλο αρχιτεκτονικό κοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τα εθνικά κοινοβούλια και τα περιφερειακά κοινοβούλια να χρησιμοποιούν πλήρως τα εφιστάμενα μέσα και πάνω απ' όλα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην κατηγορούν τις Βρυξέλλες για όλα τα στραβά του κόσμου, αλλά να κάνουν επικοδομητικές ε, προτάσεις για τη λειτουργία της Υπήρου μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προφανώς καλό όλο τον κόσμο να υπερψηφίσει αυτή την έξοχη έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ντελβό. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο.